στην εθνική νομοθεσία και να πάνε πέρα από τις ελέγξεις απαιτήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος. Κλείγενη εδώ συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Λοιπόν, κατόπιν έχουμε προφορική ερώτηση στην Επιτροπή για την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεκάστρο για πέντε λεπτά, ο οποίος είναι ο συντάκτης της ερώτησης. Κυρία Προέδρε, κύριε Επίτροπε, εξαιότιμοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια σημαντική ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε και με ευθύνη το αυξανόμενο πρόβλημα της αντίστασης στα αντιβιωτικά ε, των ζώων. Είναι θέμα στατογικό για το γεωρικό τομέα, κυρίω για το μέλλον του συστήματο τη συνοτροφία στην Ευρώπη. Τα στοιχεία δίνουν στην Ευρώπη ότι για ζωική χρήση έχουμε, δίνονται περίπου τα μισά από τα χρησιμοποιούμενα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, είναι ένα μέσο χρήσιμα που βοηθά του γεωργού να διατηρήσουν υγιή και παραγικά τα ζώα τους και να εγγυηθούν την ε, ζωή τους. Εδώ δεν είμαστε εδώ για να θεωρήσουμε ότι είναι πολύ κακό το να χρησιμοποιηθεί στη ζωοτροφία το αντιβιωτικό, αλλά να δώσει η απάντηση συγκεκριμένη η Επιτροπή για πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των φαρμάκων για να ε, μειωθεί η αντίσταση στα ζώα. Αυτό το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τη 5η Μαου του 2010 σε αυτό το πρόγραμμα δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την ε, ζωή των ζώων είχε ήδη υπογραμμίσει τη ε, διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ τη καλή ζωή των ζώων, τη υγεία του και τη δημόσια υγεία και κράτη, καλούνται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσουν με σωστό τρόπο το θέμα τη αντίσταση των ζώων στα αντιβιωτικά. Κυρίω καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει και να αναλύσει στοιχεία όσον αφορά τη χρήση όλων των προϊόντων για την υγεία των ζώων συμπεριλαμβανομένων και των αντιβιωτικών, προ σκοπό να αγγιθούμε αποτελεσματική χρήση αυτών των προϊόντων. Μετά από ένα χρόνο, η, Επιτροπή Γεωργία, τη οποία έχω τιμή να προεδρεύω, είναι εδώ για να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει όλε τι πρωτοβουλίε που θα είναι χρήσιμε για να μειωθεί αυτό το πρόβλημα το επιζήμιο που μπορεί να έχει συνέπειε και επί τη ανθρώπινη υγεία. Αυτό που πρέπει, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι να ληφθεί μια δέσμευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένη που ξεκινά, ξεκινώντα με τη στοιχεία, να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τα αποτελέσματα αυτό και να προωθήσει όχι μόνο τον έλεγχο και την έρευνα, αλλά για να εγγυηθεί καλύτερη αποτελεσματική χρήση των αντιβιωτικών, που είναι σημαντικό εργαλείο για να αντισταθούμε στι ε, ασθένειε των ζώων. Σε αυτό το μέτωπο να επιθυμίσω ότι κάποιε μελέτε καταδεικνύουν ότι μία δίαιτη ε, με χαμηλή ενεργειακή και η περιεκτικότητα ε, στα ζώα μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερε ε, ασθένειε και μεγαλύτερη χρήση των αντιβιωτικών. Σε πλήρη σεβασμό τη μέγιστη ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να απαγορευτεί ε, να χρησιμοποιηθούν τα ζωάλευρα για τα ζώα με μία κοιλιά σύμφωνα με την Επιστημονική την Ιατρική Επιτροπή τη Ευρώπη. Αυτά είναι τα αιτήματα του ψηφίσματο που θετήθηκαν στην Επιτροπή Γεωργία στι περασμένε 12 Απριλίου και θα ψηφίσουμε σε αυτή την ολομέλεια αυτό το κείμενο αύριο. Ήταν εντατική εργασία του τελευταίου μήνε και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κυρία Πόλσον, Δισέιντο και όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες για την πολύτιμη συνεισφορά τους όσον αφορά τον καθορισμό ενός κοινού κειμένου επί ενός θέματος το οποίο η διαχείριση μπορεί από τη διαχείριση αυτού του θέματο μπορεί ε, ε, να, να εξαρτάται ε, η ανταγωνιστικότητα της ζωοτροφίας στην Ευρώπη και χρειάζεται βούληση κοινή να υπάρχει συντονισμός και κοινή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο τον κύριο Άντορ. Έχετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Άντορ, δεν τον ακούνε οι διερμηνείς. Να υπογραμμίσω καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά και ανησυχεί για την απειλή για τη δημόσια υγεία που δημιουργείται από την αντίσταση κατά των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, ε, το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων να ηγηθεί στη συλλογή συγκρισίμων στοιχείων όσον αφορά την χρήση των ε, φαρμάκων κατά των μικροβίων στα ζώα, των αντιβιωτικών. Λοιπόν, έγινε η φορέας ο ΕΣΒΑΚ το τρίτο τετράμινο ε, του 2009 ξεκίνησε εργασίες του η ΕΒΑ, η ΕΜΑΚ και ξεκίνησε η προσπάθεια να αναπτυχθεί το δέον σύστημα. Τα αποτελέσματα των στοιχείων διατίθενται από 10 κράτη-μέλη, θα δημοσιευθούν τα στοιχεία των ταχύτερων δυνατών. 12 επιπλέον κράτη-μέλη εθελοντικά άρχισαν να συλλέγουν τα στοιχεία. Στόχο, διεύρυνση του συστήματο, Να καλύπτονται όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Άλλος στόχος, να έχουμε στοιχεία και περισσότερο λεπτομερή, όπως σε επίπεδο ειδών ζώων. Γιατί τα χρειαζόμαστε τα στοιχεία. Τα χρειαζόμαστε ούτω ώστε να ακολουθήσουμε προσέγγιση που θα βασίζεται επιστημονικών στοιχείων. Μόνο από αυτό το στοιχείο είναι επιστήμονε που αξιολογεί το πραγματικό κίνδυνο αυτή τη αντίσταση που οφείλεται στην χρήση αντιβιωτικών στα ζώα. Τώρα στρεφόμενος στο δεύτερο ερώτημα. Σας διαβεβαιώ, αξιότιμα μέλη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι ο έλεγχος των αναγκών στα αντιβιωτικά είναι, χρειάζεται μια πολυτομική προσέγγιση. Γι' αυτό ερχόμαστε σε επαφή με τι υπηρεσίε μα, τα κράτη-μέλη, του φορεί των κρατών μελών και άλλου εμπλεκομένου φορεί. Συνεχή επαφή υπάρχει μέσω συνεδριάσεων και δημοσίων διαβουλεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το θέμα σε στενή συνεργασία με του διάφορου αρμόδιου φορεί, κυρίω το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την πρόληψη των επιζωτιών και τον έλεγχο, την Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την Ευρωπαϊκή Οργανισμό Φαρμάκων, και το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για την ανάλυση αυτών των φαρμάκων. Και το τρίτο ερώτημα. Θέλω να πω μας αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πενταετή στρατηγική όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Θα εθετήσει ολιστική προσέγγιση και θα εμπεριέχονται συγκεκριμένε προτάσει για περαιτέρω δράση που θα πρέπει να δρομολογηθούν για να καλυφθεί το πρόβλημα αυτό για την αντίσταση στα αντιβιωτικά και για την ε, δημόσια υγεία και για τη ζωή των ε, ζώων. Θα βασιστούμε σε συστάσει και συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα ανάλογα και επί των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων που προανέφερα. Εργασίε επί τη αναθεωρήσεω των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τα σχετικά προϊόντα και τα διάφορε ζωοτροφέ με φάρμακα είναι κάτι που συνεχίζεται νέα εργαλεία και μέσα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα θα εξεταστούν εν την προετοιμασία όπως ε, την προετοιμασία για την εξολόγηση συνεπιών. Βάσει των πληροφοριών που συλλέξαμε θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των λεπτομεριών τη προτάσεω νομικού περιεχομένου που θα κάνει. Στόχο να παρουσιάσουμε στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 18 Νοεμβρίου που θα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για το 2011 για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα αντιβιωτικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Επίτροπο. Τώρα, οι ομιλητέ εξονόματο των πολιτικών ομάδων θα ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά. Η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Παύλο Δεκάστρο, τον πρόεδρο τη ε, Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων, για την πρωτοβουλία και για το προφορικό ερώτημα που έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επιτροπέ, σα άκουσα προσεκτικά να σα προσθε... σας παρακαλέσω να ξεπεράσετε την θεωρία, να περάσετε στην πρακτική, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για, για κάτι πραγματικό. Η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά, το οποίο έχει ληφθεί πολύ λίγο υπόψη τώρα σε ό,τι αφορά την εκτροφή ζώων. Χρησιμοποιούνται ε, συχνά τα αντιβιωτικά και αποτελούν ασφαλώς χρήσιμο εργαλείο, χρήσιμο μέσο για τη διατήρηση της ευημερία των ζώων. Αλλά για να είναι στη διάθεσή μας και μελλοντικά τα αντιβιωτικά ως μέσο καταπολέμησης των ασθενειών και για τα ζώα αλλά και για τους ανθρώπους χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση. Τις τελευταίες εβδομάδες στην Επιτροπή Γεωργίας ασχοληθήκαμε πολύ έντονα με το θέμα αυτό. Το συζητήσαμε πολύ έντονα και το κοινό ψήφισμα το καταθέσαμε και το υπερψηφίσαμε στις 12 Απριλίου στην Επιτροπή. Μόνο δύο ψήφοι ήταν κατά. Στριπτικό το αποτέλεσμα. Καταλήξαμε σε ένα σερωπημένο κείμενο μετά από συνεργασία με όλες τις ομάδες. Και γι' αυτό αύριο σας παρακαλώ στην ε, Σύνοβο της Ολομέλειας να το υποστηρίξουμε. Είναι ισορροπημένο το κείμενο. Λαμβάνει υπόψη την υγεία των ζώων, το θέμα της ανθεκτικότητας των αντιβιωτικών, αλλά και το θέμα της ε, διαχείρισης των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό ευχαριστώ όλους τους αρμόδιους της Επιτροπής Γεωργίας για την καλή συνεργασία και για την καλή συνύπαρξη. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και θα ήθελα να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος ε, Κάπουλα Σάντος, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συνέπειε τη χρήση αντιβιωτικών ε, για τη θεραπεία των ζωνώσεων είναι γνωστέ και, και, όλο πιο, και πιο ανησυχητικέ. Ε, ήδη ε, έχουμε απαιτητική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή θετικέ πρωτοβουλίε όπω η συλλογή πληροφοριών για την ανθεκτικότητα στην βιωτικά. Όμω όλα αυτά δεν αρκούν η Κομισιόν αναφέρθηκε σε μηχανισμούς ε, παρακολούθησης, αλλά πρέπει να υιοθετήσει και τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η συλλογή των δεδομένων να είναι πιο καθολική και πρέπει στην μελλοντική ΚΑΠ να θέσουμε και το θέμα των ορθών πρακτικών ε, ε, η ε, Επιτροπή Άγκρη παρουσίασε ένα κείμενο ε, που υποστηρίχθηκε δεόντως και θα πρέπει η Επιτροπή να το λάβει υπόψη και να το μεταφράσει ε, στην εφαρμογή μέτρων προκειμένου να έχουμε καλύτερα προϊόντα στην Ευρώπη ζωικής προέλευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ομάδα των φιλελευθέρων κυρία Πόλσεν για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Εξωτήμοι συνάδελφοι. Αυτή τη φορά κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Επιτροπή Γεωργίας. Λίγες φορές υπήρξε τόσο καλή και συνενετική συνεργασία όπως στην περίπτωση αυτή. Η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά αποτελεί πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα γιατί μας απειλεί τα μάλα. Πρόκειται για μια απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάποια στιγμή στο παρελθόν οι μολυσματικές νόσοι προκαλούσαν θανάτους στα παιδιά, στους ενηλίκους, κάποια φακτήρια προκαλούσαν πολύ μεγάλη καταστροφή και είχαμε όλοι τον ίδιο βαθμό ε, ανοσίας όμως ε, τελικά καταλήξαμε στο να χρειαζόμαστε αντιβιωτικά και κάθε φορά όσο χρησιμοποιούμε αυτά τα αντιβιωτικά χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερα και πιο ισχυρά γιατί αποδυναμώνει το νοσοποιητικό μας. Εμείς από τη σκοπιά της ε, ιατρικής προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε αν ε, υπήρχε συνολική ανθεκτικότητα. Αν δεν είχαμε τα αντιβιωτικά ως όπλο δεν θα μπορούσαμε να ε, ξεφορτωθούμε ορισμένες απειλές στην υγεία. Θα επανερχόμασταν στην εποχή των προγιαγιάδων μας και πράγματα τα οποία μας φαίνονται σήμερα πολύ απλά όπως μια οτίτιδα ε, θα μετατρέπονταν σε θανατηφόρες νόσους. Έτσι λοιπόν... Δεν ε, μπορούμε να το δούμε ελαφρά αυτό το ζήτημα, το αντίθετο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα ότι το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες σε αυτό το ψήφισμα που εγώ θα ήθελα να ε, δω εις βάθος, όμως το σημαντικό είναι εδώ να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό το θέμα της βούλησης, της ύπαρξης βούλησης να ενισχύσουμε την διαδικασία διόρθωσης ε, των ε, συνεπειών που μπορεί να προκύψουν. Εγώ αύριο θα ψηφίσω θετικά, ελπίζω όλοι να το πράξουν για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να ε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα. Για το ECR, ε, Ashworth, για δύο λεπτά. Uh, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας που έθεσε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την ανησυχία που εκφράζει σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα των, ε, στα αντιβιωτικά σε ό,τι αφορά τέτοια βακτήρια. συμφωνώ ότι θα πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει περίπτωση μεταφοράς της ανθεκτικότητας αυτής και στους ανθρώπους. Μήπως με την ανθρώπινη υγεία. Άρα υποστρίζω το σκοπό της συζήτησης και συμφωνώ ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τις διάφορες υπηρεσίες και με την φαρμακοβιομηχανία για να εκτιμήσουμε την έκταση του προβλήματος. Ωστόσο, αντίθετα με την κοινή γνώμη, δεν πρόκειται για ένα αποκλειστικό πρόβλημα που προκλήθηκε από την εντατική γεωργία. Η χρήση των αντιβιωτικών στη γεωργία ήταν σε, όλες, ε, σε όλα τα επίπεδα καλλιεργειών, μεγάλων και μικρών. Και να σας πω ότι συνήθως ε, οι μεγάλοι γεωργοί έχουν συμβατικές ε, υποχρεώσεις και ότι η προληπτική χρήση αντιβιωτικών συνήθως απαγορεύεται σε τέτοια είδους προγράμματα, αλλά είναι σαφές το εξής. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Και ανυπομονώ να ακούσω τις λεπτομέρειες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία σημεία θέλω να υπογραμμίσω. Καταρχάς, ότι θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία ορθά. Κατά δεύτερον, ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι αναλογικά. Και τρίτον, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν περαιτέρω από πλευράς κόστους και νομοθεσίας την ε, γεωργία και την ε, ιατρική. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους για δύο λεπτά. κύριος Συνάδελφοι, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για την μελλοντική εκτροφή ζώων αλλά κυρίως για την ανθρώπινη υγεία. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρόκειται για πρόβλημα της Επιτροπής Γεωργίας μόνο. Αυτό όμως που θα πρέπει να είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε απαραίτητα δεδομένα. Δεν αρκούν τα δεδομένα από 10 κρατημέλη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό πιο γρήγορα για να υπάρχει ακριβής έλεγχος. Ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι δεν έχει λάβει σωστή προσοχή είναι η εντατική εκτροφή ζώων. Θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το καταπολεμήσουμε με τη νέα γεωργική πολιτική σε ό,τι αφορά την δίκαιη εκτροφή και σωστή εκτροφή ζώων προκειμένου να τηρήσουμε και την αρχή της πρόληψης. Αυτό που χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για να μειώσουμε τέτοια περιστατικά στην γεωργία σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα. Αυτή αφορά κυρίως ε, τους εκτροφείς και τους υπαλλήλους τους. Και αυτό που προκαλεί ανησυχία στο πλαίσιο αυτό είναι το εξής. Υπάρχει υποψία ότι υπάρχει και ανθεκτικότητα η οποία αναπτύσσεται μέσα από τα τρόφιμα και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε ό,τι αφορά την υγεία του Ευρωπαίου πολίτη στην τελική ανάλυση. Κατεπικόντως λοιπόν πρέπει να δράσουμε και το ότι το 50% των αντιβιωτικών χρησιμοποιείται για την εκτροφή των ζώων είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί στο να καταλήξουμε ότι πραγματικά είναι υπερβολικά το ποσοστό αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο στους επόμενους γεγραμμένους. Καταρχήν Νικολέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η Παγκοσμία Μέρα Υγείας στις 7 Απριλίου είχε ε, ως θέμα την ολθεκτικότητα στα αντιβατικά ως παγκοσμία πύλη στη δημοσία υγεία. Στην Ευρώπη 27.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά. Ε, τροφές ζωικής προέλευσης μπορεί να είναι ε, ο λόγος αυτής της ανθεκτικότητας γι' αυτό το θέμα που συζητούμε σήμερα είναι άκρο σημαντικό εδώ η πιο σημαντική λέξη είναι να, ε, η σοφροσύνη, δηλαδή δεν είναι τα αντιβιωτικά που είναι κακά, ε, αλλά η χρήση που τους γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά με σοφροσύνη και για τους ανθρώπους και για τα ζώα η πρόταση αυτού του ψηφίσματος να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ό,τι αφορά τώρα ε, τα αντιβιωτικά και τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές. Ε, αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει διεθνή συμφωνία. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν το 50% του κρέατος που τέθηκε σε δοκιμές συμπεριλαμβάνουν οι βακτήρια που αντιστέκονται σε ε, τρία είδη αντιβιωτικών. Εγώ πρέπει να πω ότι οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι έχουν κουραστεί να είναι οι μόνοι που ακολουθούν τους κανόνες ε, και χάνουν χρήματα από αυτό. Ευχαριστώ, Ρόντους, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ε, αποτρέψουμε περαιτέρω ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνους ε, σε ό,τι αφορά την χρήση αντιβιωτικών στην υγεία των ανθρώπων. Ε, αυτή επηρεάζεται και από την χρήση αντιβιωτικών για τα ζώα. Θα πρέπει αποφασιστικά να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πεθαίνουν κάθε χρόνο 25.000 άνθρωποι λόγω ανθεκτικών βακτηρίων. Θα πρέπει προληπτικά να ληφθούν μέτρα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη-μέλη ε, γίνεται ευσυνείδητη χρήση των αντιβιωτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εκτροφή των ζώων να γίνουν όλες οι προσπάθειες προκειμένου να διατηρούνται υγιή τα ζώα από τη γέννησή τους μέχρι την ενήλικη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι και το α και το ω για την ε, αποτροπή χρήσης αντιβιωτικών. Και εδώ είναι σημαντική η ζωοτροφή. Αλλά είναι σημαντική η εκτροφή των ζώων. Θα πρέπει ανοιχτά να μιλήσουμε για εναλλακτικέ μεθόδους, όπως ε, τη χρήση ομοιοπαθητικών ε, φαρμάκων στην ζωοτροφή στην εκτροφή ζώων. Χρειάζεται προ αυτήν την κατεύθυνση πιο πολύ γνώση, πιο πολύ έρευνα. Σας ευχαριστώ. Γερμπράντι, για μισή λεπτό. Κύριε Γερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επιτροπέ, συνάδελφοι. Η χώρα μου, η Ολλανδία, είναι πρωταθλητή στον κόσμο. Όχι στο ποδόσφαιρο, δυστυχώ το χάσαμε το πρωτάθλημα την προηγούμενο χρόνο, αλλά στη χρήση αντιβιωτικών σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία. Καμία χώρα δεν χρησιμοποιεί τόσο, πολύ, τόσο πολλά αντιβιωτικά στην κτηνοτροφία. Και αυτό έχει μεγάλε συνέπειε, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 25.000 άτομα πεθαίνουν από βακτηριακές μολύνσεις. Αυτό περνάει μέσα από τα τρόφιμα. 90% των κοτόπουλων, του κρέας κοτόπουλου, περιλαμβάνει ανθεκτικότητα σε βακτήρια. Και ακόμα και σε λαχανικά βρέθηκαν τέτοια αντιβιωτικά, τα οποία ε, περνάνε μέσα από το χώμα. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό, Πρόεδρε, με αυστηρά μέτρα θα πρέπει να περάσει η χρήση λιγότερων αντιβιωτικών και να αποδείξουμε ότι μπορεί να είναι ε, υγιής ο κλάδος της κτηνοτροφίας. Το είπε και ο Επίτροπος ότι τον Νοέμβριο θα υποβάλει σχετικά μέτρα. Το 2012 θα υπάρξουν και συγκεκριμένες προτάσεις να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει καταπήγοντα χαρακτήρα στο θέμα αυτό. Να μην εξαρτηθεί από τα κράτη-μέλη τα οποία είναι υπερβολικά αργά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σωστών μέτρων. Σα ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη διαδικασία προσέγγιση προσοχή τη Προέδρου με την κυρία Μαγκίνε που έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σαφέ ότι υπάρχει γενική ανησυχία όσον αφορά τα αντίσταση στα αντιβιωτικά από τα διάφορα κόμματα. Όμω μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε στοιχεία από 10 κράτη-μέλη και δεν τα έχουμε ακόμα στη διάθεσή μα. Μιλάμε για ανησυχίε οι οποίε δεν είναι ε, λεπτομερή στοιχεία και χρειαζόμαστε πληροφορίε. Θα ήθελα να δω έναν πίνακα κρατών μελών πώ χρησιμοποιούν τα φάρμακα αναπληθισμό ζώων για να μπορέσουμε να δούμε ποιε χώρε ακολουθούν την καλύτερη πρακτική για να τι βαθολογήσουμε έναντι άλλων που δεν κινούνται σωστά. Όχι για να δαχτυλοδείξουμε, αλλά για να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη που ίσω χρησιμοποιούν υπερβολικά τα αντιβιωτικά να βελτιώσουν τι πρακτικέ του στι κτηνιατρικέ. Και είναι σωστό να πούμε στη συζήτηση ότι δεν χρησιμοποιούν τυχαία τα φάρμακα οι κτηνοτρόφοι όταν αρρωσταίνουν τα ζώα τα χρησιμοποιούν γιατί είναι και ακριβά τα αντιβιωτικά δεν τα χρησιμοποιούν έτσι τυχαία σαν όπως θα πότιζαν νερό τα ζώα του. Χρειάζεται ισορροπημένη συζήτηση. Α πάρουμε τι πληροφορίες, περιμένουμε να δούμε τη στρατηγική τον Νοέμβριο, ούτω ώστε να μην έχουμε αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα ζώα μας και για τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Γιάρ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Χαίρομαι που το θέμα αυτό συζητείται. Η χρήση των ε, αντιβιωτικών στα, στην κλινιοτροφία έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθεί η υγεία των ζώων, αλλά αν χρησιμοποιηθούν ε, υπερβολικά δημιουργείται κίνδυνο και για του ανθρώπου. Άρα χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση που θα εδράζεται επιστημονικών δεδομένων. Διότι η χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη στο μέλλον. Τούτων λεχθέντων θα πρέπει να υπερασπιστούμε την υγεία των ανθρωπίνων όντων. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πρόταση της εκθέσεως είναι έξοχη και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προτάση μάλλον του Κοινοβουλίου που έγιναν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να ληφθούν υπόψη. Είναι καλέ προτάσει. Κυρίω πρέπει να γίνει ανάλυση τη καταστάσεω όλα τα κράτη-μέλη προ όφελο των ζώων τη Γεωργία, τη Ευρωπαϊκή και πάνω απ' όλα προ όφελο των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και τώρα δούμε το λόγο στον κύριο Μικολαζίκ. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. να υποδείξω το εξής. Κάτι κοινό στην ε, υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων και ζωών σε όλα τα μικροβιολογικά συνέδρια όταν μιλάμε για την ε, ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά στους ανθρώπους μιλάμε για τον σταφυλόκοκο και την ανθεκτικότητα σε αυτούς τους ε, σε αυτές τις μολύνσεις δεν υπάρχει πλέον αντιβιωτικό το οποίο θα ήταν αποτελεσματικό σε τέτοια περίπτωση. Πώς καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση από την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών, των αντιβιωτικών, στην εκτροφή ζώων. Προληπτικά χορηγούνται μέσω των ζωοτροφών στα ζώα τα αντιβιωτικά αυτό. Και ως εκ τούτου προκύπτει ανθεκτικότητα και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ε, προστατευτούν από μολύνσεις τις οποίες κολλάνε στα νοσοκομεία, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξει δεδομένα και να αναζητήσει, να υποστηρίξει μάλλον την αναζήτηση νέων αντιβιωτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Ευχαριστώ Πάσκα. Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Η χρήση προϊόντων της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας στα τρόφιμα αποτελεί την οδό μέσω της οποίας καταλήγουν τα φάρμακα αυτά στον ανθρώπινο οργανισμό. Η χρήση της σύγχρονης χημίας και της φαρμακευτικής στον τομέα τον αγροτικό θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση του αντικτύπου για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες και για την ανθρώπινη ζωή. Η προληπτική αυτή χρήση, μάλλον η προληπτική αυτή εξέταση θα μας αποκαλύψει τις νέες δυνατότητες σε ό,τι αφορά και τις νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για έναν ενδυνάμει κίνδυνο η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Αλλά πρόκειται για ένα πολύ σύμφωτο θέμα και έτσι θα πρέπει να το θεωρήσουμε. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Άντορ, παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η στρατηγική τη Κομισιόν για την ανθεκτικότητα στα ιδιωτικά, παρουσιάστηκε το Νοέμβριο. Ε, θα έχουμε και περαιτέρω ιδέε για το πώ η Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη και τους stakeholders μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της ανθεκτικότητας στα ιδιωτικά σε όλου του τομεί. Μπορεί να χρειαστούν κάποιε αλλαγέ στην νομοθεσία, αλλά σε ορισμένους τομείς, ίσως όχι. Πρέπει να επιλέξουμε το σωστό εργαλείο για το κάθε ε, τομέα συμφωνώ ότι αυτό δεν αποτελεί ένα θέμα αποκλειστικά κτηνοτροφίας ε, γι' αυτό θέλουμε να περιορίσουμε την ε, ανθεκτικότητα ε, στα αντιβιωτικά ε, την αντικομικοβιακή ανθεκτικότητα υπάρχουν διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης κτλ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ε, πρέπει να συλλέξουμε τα στοιχεία για να έχουμε καλύτερη κατανόηση του φαινομένου. Τα κράτη-μέλη δείχνουν ενδιαφέρον να παράσχουν δεδομένα και αυτό είναι θετικό. Και ναι, έχουμε το χρονοδιάγραμμα για δράση. Προπαρασκευαστικό έργο συνεχίζονται, αναθεώρηση των κανόνων ε, για τα εκτενιατρικά φάρμακα νομοθετικές προτάσεις ε, θα έλθουν θα καταφτάσουν το 2012. Η Κομισιόν καλωσορίζει την πολύτιμη συνεισφορά του Κοινοβουλίου και περιμένει να συνεχίσει τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους από όλους τους τομείς με τον κοινό στόχο να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος, λίγη εδώ συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση αύριο 12 Μαΐου